Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na popołudniowym spotkaniu komisji. Καλώς ορίσατε στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Για σήμερα το απόγευμα έχουμε να ασχοληθούμε με το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Καλωσορίζω τους ομιλητές μας, για την απόψινή συνεδρίαση. από την ΕΣΟ, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, από το Πανεπιστήμιο της ε, Κρακοβίας, την κυρία Ρουντέλη επίσης από τον κλάδο βιομηχανία, handlung επίσης, από τα συνδικάτα οικοδόμων και επίσης θα ήθελα να, καθ... καλωσορίσω την κυρία Άγνες Γιανκέριους που εκπροσωπεί ένα συνδικάτο από την Ολλανδία. Καλώς ορίσατε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε δύο ώρες στη διάθεσή μας και θα ήθελα να ζητήσω από τους εμπειρογνώμονες να μιλήσουν για έξι λεπτά. Λυπάμαι, αλλά αυτοί οι κανόνες μας. Να ξεκινήσω λοιπόν τον πρώτο εμπειρογνώμονα, Λίνα Κάρ, από το ETU. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας στην Επιτροπή Απασχόλησης για το ETUC Είχαμε εδώ και καιρό ζητήσει την αθεώρηση οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Για μας αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2007 με 2008. Λαβάλ Κομισιόν κατά Λουξεμβούργου. Είχαμε αυτή την υπόθεση. Και είχαμε τέσσερις αποφάσεις που αφορούσαν την νέα αγορά και την κοινωνική Ευρώπη. Δυστυχώς, η κοινωνική Ευρώπη κατά την άποψή μα έχασε τότε την υπόθεση. Η κοινωνική Ευρώπη και οι απασχολούμενοι συγκεκριμένα ήταν χαμένοι αυτή τη διαμάχης. Πριν αυτές τις τέσσερις υποθέσεις η ερμηνεία ήταν διαφορετική. Δηλαδή η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων αποτελούσε ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία των εργαζομένων όσον αφορά την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, όμως έχει μετατραπεί πια σε ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει την παροχή των υπηρεσιών αλλά δεν προστατεύει καθόλου πια τους εργαζόμενους. Έχει γίνει η ζημιά και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε εδώ και χρόνια την αναθεώρηση της οδηγίας και χαιρόμαστε που βρίσκεται πια μπροστά μας η αναθεώρηση. Εν τω μεταξύ, η αναθεώρηση του 96 γι' του 14 για αυτήν είχαμε την εκτελεστική οδηγία και η μεταφορά εξέπνευσε τον Ιούνιο φέτος. Ξέρουμε ότι κάποιες χώρες ε, έχουν καθυστερήσει, δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία ακόμα και πριν την αναθεώρηση της οδηγίας είχαμε ήδη συζητήσεις και ακούγαμε διάφορα επιχειρήματα. Παρ' όλα αυτά, η τωρινή αναθεώρηση αφορά τελείως διαφορετικά θέματα που δεν σχετίζονται. Βεβαίως μας ενδιαφέρουν οι γρήγορες μεταφορές της οδηγίας γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν καταχρηστικές αποσπάσεις που οδηγούν στην εκμετάλλευση εργαζομένων. Και σήμερα το πρωί συζητούσαμε με Πολωνούς από τα ταχυδρομεία και μας και ε, αποσπασμένους και μας έλεγαν κάποιες ιστορίες αρκετά ανησυχητικέ. Ελπίζουμε επίσης να αποφύγει αυτό το φαινόμενο θηρίδας η οδηγία και να υπάρχει μια πραγματική σχέση με την χώρα προέλευσης. Ελπίζουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά κάποιες ε, καταχρήσεις όσον αφορά την υπεργολαβία και θα πρέπει βεβαίως να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Η αναθεώρηση πάντως εξετάζει διάφορα ζητήματα και διαφορετικά. Νομίζω ότι ένα από τα κυριότερα θέματα εδώ που θα πρέπει να κοιτάξουμε στα πλαίσια της οδηγίας 96 είναι το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει έντονο ανταγωνισμό διασυνοριακά εις βάρος των εργαζομένων και τη ίση μεταχείριση των εργαζομένων στον χώρο εργασία. Επίσης, έχω και ένα ερώτημα προς όλους σας και προς τους εργοδότες. Όπως το βλέπω εγώ, εδώ έχουμε και άνισο ανταγωνισμό, αθέμητο ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις, για του εργοδότε. Επίση, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι οι εργάτες δεν είναι ένα αγαθό, δεν είναι ένα εμπόρευμα. Δεν το αγοράζουμε και το πουλάμε. Και όπως σας έλεγα προηγουμένως, καλωσορίζουμε και χαιρετίζουμε την αναθεώρηση οδηγίας. Βεβαίως υπάρχουν κάποια ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν περαιτέρω, δηλαδή το θέμα των αμοιβών. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι ευρύτερο και αντανακλά στην ουσία το όλο ζήτημα των αμοιβών των απασχολουμένων σε όλες τις χώρες μέλη. Τώρα, αν ο ελάχιστο μισθό ή ελάχιστη αμοιβή αποτελεί ρομή για την εργασία, θεωρώ ότι ξεκάθαρα η απάντηση είναι αρνητική. Οπότε και αυτό θα πρέπει να το δούμε στα πλαίσια τη αναθεώρηση τη οδηγία σήμερα. Επίση, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το θέμα της αμοιβή των εργαζομένων είναι εθνική αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Για μας η επίτευξη ίσης αμοιβή, δίκαιης αμοιβή είναι θέμα αρμοδιότητας, γιατί η ανθεώρηση βεβαίω ασχολείται με τα θέματα των συλλογικών συμβάσεων και παραβλέπει άλλα ζητήματα. Θεωρούμε ότι η διετία ως περίοδος απόσπασης είναι πολύ μεγάλη και θεωρούμε ότι είναι αντικείμενο κατάχρησης η Πρόεδρος. Ε, σας παρακαλώ ολοκληρώστε. Θα έπρεπε λοιπόν να διευρύνουμε την μικρή βάση το κεφάλαιο της κοινωνικής πολιτικής και θα πρέπει να σεβαστούμε την ανεξαρτησία των εταίρων. Και θα πρέπει να δούμε ακριβώ και τι γίνεται και με την υπεργολαβία, όπου έχουμε πολλά αρνητικά φαινόμενα. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα προσκαλέσατε. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο. Νέλη Στράμπε από την ομάδα εργασία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Προτού αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, που θα συνεισφέρουν στη δουλειά σας. Ορισμένες γενικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν βλέπουμε να χρειάζεται ανάγκη να θεώρηση οδηγία. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τους αφαρμοστέους κανόνες στο μέλλον. Διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία, διότι δεν έχει εφαρμοστεί σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και η εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων ελέγχου, πιστεύουμε, καθυστερεί. Γι' αυτό χαιρετίζουμε το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη τη ορθή εφαρμογή και ταχής εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Και πιστεύουμε ότι πολλέ από τι παράτυπε περιπτώσει που ακούμε και ε, αντιπροσωπεύουν τις νομικές εταιρείες, πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία τα προβλήματα αυτά οφείλουν στο γεγονό ότι δεν έχει εφαρμοστεί ορθά η οδηγία και πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι συμφωνήθηκε αυτή η οδηγία το 1996 από όλα τα κράτη-μέλη εν ώψη της διεύρυνσης και ως αντικείμενο είχε να δημιουργήσει ένα παιχνίδι ένα πεδίο με παιχνίδι ισονόρους, όρους, ε, κυρίως λόγω των θετικών επιπτώσεων της ενιαίας αγοράς. Και το, το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ο, ο Επίτροπος στην Κρακοβία είπε ότι χρειάζονται διασυνοριακές υπηρεσίες που έχουν ως άξονα την εξειδικευμένη εργασία και τις ικανότητες, όπως και από τις διαφορές ε, στο κόστος εργασίας. Συμφωνούμε, διότι γνωρίζοντας ε, ποια είναι η επιπλέον δαπάνη με την απόσπαση ενός εργαζόμενου, είναι εκείνο το οποίο θα καθορίσει τις αποσπάσεις είναι οι ειδικότητε και αρμοδιότητες. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη ότι η, από όλα τα κράτη-μέλη και εργαζομένων μπορεί να καλύψει τα κενά στις ειδικότητε. Πάντοτε παραμένοντας μέσα στα νομικά πλαίσια της χώρας προέλευσης. Το θέμα έχει γίνει ένα θέμα Ανατολής και Δύσης. Αυτό είναι λάθος πιστεύω μετά από την Πολωνία είναι η Γερμανία και η Γαλλία οι χώρες ε, που έχουν ε, αποσπασμένους εργαζόμενους και έχουν ένα μεγάλο ποσοστό, ένα μεγάλο ποσοστό αποσπασμένων εργαζομένων ετησίως. Κατόπιν στη τρίτη και τέταρτη σειρά έρχεται η Ολλανδία και η Ισπανία. Δεν είναι ανατολικέ χώρες, είναι δυτικέ χώρε και χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα απόσπασης εργαζομένων. Επίσης, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον τομέα των οικοδομών. Το ξέρω ότι ο οργανισμός, ε, η Ομοσπονδία ε, των Οικοδόμων και των Εργατών Ξύλου δεν έχει προσκληθεί, αλλά παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί, σας, μαζί τους για να μάθετε τι συμβαίνει στον κλάδο των οικοδομών. Τώρα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο περιορισμός των αποσπάσεων σε 24 μήνες. Αυτός είναι ένας νέος κανόνας. Και τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν μια γερμανική εταιρεία στείλει έναν εργαζόμενο στη Γαλλία, αυτός ο αποσπασμένος θα πρέπει να αλλάξει τη σύμβασή του με σύμβαση ε, γαλλικού δικαίου. Και όταν επανέλθει στη Γερμανία πάλι θα πρέπει να εμπίπτει στη σύμβαση του γερμανικού δικαίου. Αυτό δεν είναι καλό πιστεύουμε ούτε για την εταιρεία ούτε για τον υπάλληλο. Στην πρόταση της Επιτροπής μόνον εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει παρέκκληση με μονομένες συμφωνίες μπορεί κανεί να, μείνει, ε, να παραμείνει με τη σύμβαση της χώρας προέλευση. Και σε ειδικέ περιπτώσεις μόνον αυτό θα επιτραπεί. Συνεπώς δεν πρέπει αυτή να είναι πραγματική δυνατότητα ε, για τις εταιρείες και για τους απασχολούμενους. Επίσης, ε, δεν πρέπει να προσθέτει κανείς θέσεις απόσπασης που επαναλαμβάνονται διότι πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν μιλάμε μόνο για τον κλάδο των οικοδομών και για υπεργολαβίες. Η οδηγία αφορά επίσης ε, τα άτομα που μεταφέρονται μέσα σε μια επιχείρηση και χρησιμοποιούνται επαναλημμένες αποσπάσεις. Για παράδειγμα, πολλές εταιρείες ευτυχώς έχουν προγράμματα εκπαίδευσης για νέους που κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες Ευρώπης και η πρόταση της Κομισιόν ε, σημαίνει ότι σε δύο χρόνια θα πρέπει ε, αυτό το άτομο που μετατίθεται ε, να εμπίπνει σε διαφορετικές νομοθεσίες ανάλογα με την απόσπασή του. Σίγουρα έτσι νέοι ε, βλέπουν πόσο περίπλοκη είναι η Ευρώπη με την περίπλοκη εργατική νομοθεσία ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Επίσης, η ελάχιστη αμοιβή ε, δεν θα αναφερθώ εκεί, η συνάδελφος θα αναφερθεί, όσον αφορά τις υπεργολαβίες. Η πρώτη επιτροπή σημαίνει ότι ο υπεργολάβος πρέπει να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τους κανόνες της χώρας υποδοχής, το οποίο σημαίνει ότι κάθε φορά ότι ο εργοδότης αλλάζει υπεργολάβο, τότε οι υπάλληλοι επίσης εκ του νόμου θα αλλάξουν ε, συνθήκες πληρωμής, αμοιβή δηλαδή και εργασία. Κάθε φορά δηλαδή ότι ο εργολάβος, ο εργοδότης αλλάζει, αλλάζουν και οι, οι όροι εργασία και αμοιβή του εργαζόμενου. Δεν είναι όμως σωστό. Θα πρέπει οι συνθήκες αμοιβή και εργασία για τον εργαζόμενο να παραμένουν αναλύωτες. Δεύτερον, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείε θα πρέπει να κάνουν διάκριση. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Ναι, το συμπέρασμα είναι ότι αυτό τελικά είναι ε, είναι ένας εφιάλτης για τις εταιρείε. θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας, ελπίζω με τις απαντήσεις να δώσω και άλλα παραδείγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ακή Εβανχόκ. Σίγουρα δεν ε, έχω προφέρει σωστά το όνομά σας, ζητώ συγγνώμη. Καθηγήτρια ιδιωτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Έχετε το λόγο. Okay, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να σχολιάσω το θέμα αυτό. Εγώ είμαι καθηγήτρια, θα μιλήσω λοιπόν ε, λίγο πιο θεωρητικά όσον αφορά τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα αυτών των κανόνων και της νομοθεσίας από το θέμα της ελάχιστης αποδοχής, του ελάχιστου μισθού θα ξεκινήσω. Είναι κάτι που σίγουρα βασίζεται στην υπάρχουσα κατάσταση. Υπάρχουν ε, τα κατώτατα όρια αποδοχών σε πολλές χώρες. Εγώ είμαι και δικαστής σε εμπορικές υποθέσεις ε, στην ε, Ολλανδία και αυτό που πάντα ε, εξετάζουμε είναι να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ποιο είναι το πραγματικό ωριο μισθολόγιο ή ημερομίστιο που δίνουν στους εργαζόμενους. Και βεβαίως αυτά δεν καθορίζονται πάντα από την νομοθεσία. Γι' αυτό και θα πρέπει να αφαιθεί ε, χώρος στους κοινωνικούς εταίρους, στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, στις επιχειρήσεις για να γίνει διαπραγμάτευση και να οριστούν αυτά τα επίπεδα αποδοχών. Αυτό που προβλέπει ο νόμος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει διαπραγμάτευση και οι κοινωνικοί εταίροι αφού συνάψουν μία συλλογική σύμβαση, αυτή να ισχύει και να καλύπτει όλον τον ε, κλάδο. Και το θέμα είναι αν ε, θέλουμε να ε, παίξουν αυτό το ρόλο οι κοινωνικοί εταίροι ή να τον αφήσουμε στον κράτος. Η πρόταση που ε, εξετάζουμε σήμερα δυστυχώς αποδυναμώνει λίγο την σημερινή αρμοδιότητα και ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Βεβαίως οι κοινωνικοί εταίροι σήμερα ε, λειτουργούν στα συστήματα που υπάρχουν και επιβάλλονται οι κανόνες τους αφού βεβαίως ε, υπογραφούν συλλογικές ε, συμβάσεις και στις εταιρείε που αναλαμβάνουν την υπεργολαβία. Δυστυχώς βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις. Το θέμα παραδείγματος χάρη της μετερικής απασχόλησης, των ε, εταιριών Τις εταιρείες λοιπόν που τοποθετούν ε, υπαλλήλου ε, με μερική απασχόληση σε κάποιες εταιρείες. Και πολλές φορές βλέπουμε οι εξαιρέσεις αυτές να μην ε, υπόκεινται σε καμία από τις ε, εργατικές νομοθεσίες ή πρακτικές ή συλλογικέ συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για τον ε, κλάδο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι μηχανισμοί, όλοι αυτοί οι κανονισμοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τις περιπτώσεις αυτές, όλο τον ιδιωτικό τομέα, το θέμα τώρα της διετίας. Έχω πολλά να πω γι' αυτό. Γιατί εδώ βεβαίως ε, υπάρχει και η προϋπάρχουσα νομοθεσία και είδα πολλές αντιφατικές δηλώσεις στην πρόταση και βεβαίως δεν ε, εκπλήσωμαι γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή η πρόταση θα είναι αποτελεσματική. Μετά από δύο χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει η τοποθέτηση του εργαζομένου, η έδρα του, άρα σε αυτή την περίπτωση είναι λογικό να ισχύει η νομοθεσία του κράτους το οποίο δραστηριοποιείται. Αλλά αν χωρίς να έχει αλλάξει η τοποθεσία στην οποία ζει και εργάζεται ο εργαζόμενος αν έτσι και αλλιώς αλλάξει η νομοθεσία, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ισχύει το σύνολο των κανόνων αυτής της νομοθεσίας και για τις απολύσεις και για τις αποδοχές θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να αλλάξει όλο το φάσμα των διατάξεων και των νόμων που ε, ισχύουν. Έχω ένα λεπτό στη διαθεσή μου, 40 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας ότι για την περίπτωση έτσι όπως την εξετάζουμε για τους αποσπασμένους εργαζόμενους αυξάνεται ο κίνδυνος εάν δεν είναι σαφές ποια είναι η προστασία και ποια είναι η νομοθεσία στην οποία υπόκειται ο εργαζόμενος. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπόκεινται στην νομοθεσία και στους ισχύοντες κανόνες της απόσπασης στην χώρα από την οποία προέρχονται και πιστεύω ότι στην περίπτωση τουλάχιστον των ε, δικαστηρίων στα οποία μπορεί να προσφύγει ο εργαζόμενος αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και ελπίζω ε, να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Τήρησα το χρόνο μιλίας μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος ο κύριος Μάρεκ Μπανιό από το Πανεπιστήμιο της ε, Κρακοβίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Κυρίες και κύριοι, κύριοι και κύριες βουλευτές, ευχαριστώ πολύ. Και είμαι ερευνητή, πρέπει να σας πω, και αναζητώ τους λόγους ύπαρξης αυτής της πρώτης οδηγίας. Εμείς εδώ στην Ένωσή μας θεωρούμε ότι η εργασία θα πρέπει να αμείβεται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το είπε ο Ζαν Κλοντ σε μια μιλία του το 2014. Δεν έχουμε να κάνουμε με την δίκαιη αμοιβή ή ίση αμοιβή, αλλά ίσους τρόπους υπολογισμού της αμοιβή και ουσία έχουμε κάνει με τους ίσους όρους υπολογισμούς και όχι εξίσωση τη αμοιβή. Ήθελα να το καταστήσω αυτό σαφέ από την αρχή, γιατί κάτι άλλο που λέγεται για την οδηγία αυτή είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερες αποσπάσεις, όχι λιγότερε αυτό το είπε η Επίτροπο κυρία Τάισεν. Και εδώ στην πρόταση βλέπουμε ότι ποιος είναι αυτός ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό, κάνοντας αποσπάσεις πιο περίπλοκες και ακριβές και περιορίζοντάς τις χρονικά. Αυτό για μένα είναι κάπως παράδοξο ως ε, ερευνητή. Και έχουμε και αυτά που είπε η κυρία Τάισεν για μια ισότιμη μεταχείριση. Ωραία, ισότιμη μεταχείριση. Αλλά ε, πρέπει να ξέρουμε για ποιους δυσκολεύουν τα πράγματα. Οι τοπικέ επιχειρήσει, επιχειρήσει που κάνουν αποσπάσει, οι εργαζόμενοι, για ποιου. Έκανα λοιπόν μια έρευνα έτσι, ταπεινή δικιά μου προσωπική και λάβαμε 16 απαντήσεις. Ξέρω δεν είναι εντυπωσιακό ο αριθμός, αλλά σε αυτές τις 16 ερωτήσεις καλύψαμε 20.623 έγγραφα α1. Πάνω από 20.000 λοιπόν περιπτώσεις αποσπάσεων και αν χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ συντηρητικό περιορισμό ή ένα ορισμό υπολογισμό αυτόν τον Α1 ανά υπάλληλο, μιλάμε για 15-16.000 ε, αποσπασμένους υπαλλήλους την τελευταία τριετία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότερες αποσπάσεις αφορούν τη Γερμανία όπου στα δύο πρώτα χρόνια της ε, έρευνας δεν είχαμε την εφαρμογή του κανονισμού του ελάχιστου μισθού, του κατώτατου μισθού. Η δομή λοιπόν του κόστου, της απόσπασης των εργαζομένων του εργατικού κόστους σχετικά με την έρευνά μας είναι ότι τα στοιχεία μας προέρχονται από πραγματικά δομένα από τα βιβλία των επιχειρήσεων που έλαβαν τα ερωτηματολόγια το οποίο ως θεματολόγιο είναι υψηλής ποιότητας. Γιατί αυτές ακριβώς είναι επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν, μάλλον υπέστησαν τους ελέγχους τοπικών αρχών και επιβίωσαν. Τώρα, τα αρνητικά αυτή τη έρευνα είναι ότι καλύπτονται μόνο λίγε επιχειρήσει και υπάρχει ένα είδο έτσι σχεδόν αυθαίρετη επιλογή. Αλλά συνεχίζω και ξαναλέω ότι έχουμε να κάνουμε με πάνω από 20.000 Α1. Είχαμε λοιπόν αποσπάσεις σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο. Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτό. Τώρα για τους κλάδους των αποσπάσεων, οικοδομή, οι περισσότερες, φροντίδα ηλικιωμένων, παραγωγή, επιμελητεία, συντηρουργία και τα πρώτα ευρήματα της έρευνας αυτής ήταν ότι το χαμηλότερο καθαρό εισόδημα ήταν 5,98 καθαρά την ώρα προφόρων. Όλα, συγγνώμη, μεταφόρους. Αν όμως δούμε μεικτά, φτάνουμε στα 10 ευρώ. 9,97 συγκεκριμένα. 15-16% παραπάνω από τον ελάχιστο μισθό. Οπότε εδώ η πρώτη αντίληψη καταπίπτει ότι βασίζεται ακριβώς σε φθηνά εργατικά χέρια η απόσπαση. Όχι. Φαίνεται ότι πληρώνονται λίγο παραπάνω, 15-16% από τον κατώτατο μισθό. Αλλά λίγο χαμηλότερο από το περίπου μέσο όρο των αμοιβών στις χώρες της απόσπασης. Αυτό είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν κάποια κόστη εργασίας, τα οποία σχετίζονται μόνο και αποκλειστικά με το γεγονός ότι αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε μια άλλη χώρα μέλος. Αυτά είναι τα κόστη που αντιμετωπίζουν οι χώρες όταν περνάνε τα σύνορα, τη στιγμή που υποτίθεται δεν έχουμε σύνορα. Όσον αφορά λοιπόν τους καθαρούς μισθούς, εισφορές κλπ υπάρχουν κάποια κόστη τα οποία θα λέγαμε ότι είναι διασυνοριακά μαζί με τα πάγια κόστη και τα μεταβλητά κόστη τα οποία σχετίζονται μόνο με την διασυνοριακή μετα... μετακίνηση, δηλαδή ταξίδι, κατάλημα κλπ. Εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται ακριβώ και με το βάρο για τι ε, τοπικέ επιχειρήσει. Α πούμε, έχουμε ένα κόστο μετάφραση, κόστο επιθεωρησιακή ε, ε, ε εργασία, ε, κόστο για την λήψη εγγράφων Α1. Αυτά είναι κόστη τα οποία οι επιχειρήσει δεν θα καλύψουν. Το συμπέρασμα λοιπόν ότι αυτά τα επιπλέον κόστη ανέρχονται στο 29% του συνολικού κόστους εργασίας. Το οποίο σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν αποσπάσεις αντιμετωπίζουν συμπληρωματικά κόστη τα οποία οι τοπικές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση αλλά και για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ την κυρία Ρουμπέλη, πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαίων Εργοδοτών εξ ονόματος ε, της ε, βιομηχανίας μετάλλων, μηχανουργίας και τεχνολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω προκαταρκτικές παρατηρήσεις ε, προτού εισέλθω προς το κέντρο του θέματος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η απόσπαση εργαζομένων συνδέεται στενά με την ανάπτυξη του εμπορίου και των επιχειρήσεων και είναι απαραίτητη η απόσπαση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως στον κλάδο μας. Η βιομηχανία ε, των μετάλλων και μηχανουργίας και τεχνολογίας αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ανταγωνισμό διεθνώς και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, διότι διαφοροποιείται από τους άλλους κλάδους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις μας, πολλές από αυτές, ακόμα και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεταθέτουν, αποσπούν, ε, ε, οι εργαζόμενους που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε επειδή εξάγουν προϊόντα, αλλά επίσης εξάγουν και υπηρεσίες, όταν δηλαδή κάνουν εκπαίδευση, συντήρηση, επισκευή μηχανημάτων ή στα πλαίσια ε, της ε, κινητικότητας, ενδο, της ενδομιλικής κινητικότητας. Επειδή μιλάμε για κοινωνικό dumping, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εάν ο κλάδος μας αποσπά εργαζόμενους είναι επειδή δεν έχουμε αρκετούς εξειδικευμένους εργαζόμενους. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να έχετε υπόψη όταν συζητήσετε αυτή την πρόταση για την απόσπαση. Εάν λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι αποσπασμένοι ή αν χρειάζεται να αποσπαστούν επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες σε πολλές χώρες. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αποσπασμένους είναι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Βεβαίως, σε άλλου τομεί, ε, στον οικοδομικό, στη γεωργία, στι μεταφορές, υπάρχουν προβλήματα, το γνωρίζουμε αλλά συνδέονται περισσότερο σε καταχρήσει, σε ατασταλίε, σε μη εφαρμογή τη υφιστάμενη νομοθεσία και εκτιμούμε το γεγονό ότι πρέπει να βρεθούν λύσει στα προβλήματα. Είμαστε κατά τις παράνομη εργασία όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα είναι και εμεί, οπωσδήποτε είμαστε κατά τι παράνομη εργασία, Αλλά δεν δεχόμαστε και την ιδέα ότι για να λύσουμε ορισμένα προβλήματα ότι, αυτή, δηλαδή, ότι είναι μια λύση η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Διότι θα δημιουργηθούν προβλήματα σε εκείνους που δεν έχουν προβλήματα. Στον κλάδο μας δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα. Και έχουμε την εντύπωση ότι με την αναθεώρηση αυτή τη οδηγία δημιουργείται προβλήματα για όλες τις εταιρείες μέλη. Και μα είναι δύσκολο να δεχθούμε αυτή την πρόταση, διότι αν ορισμένοι κλάδοι έχουν προβλήματα, τότε πρέπει να βρούμε λύσεις προσαρμοσμένες σε αυτά τα προβλήματα. Βεβαίω, Πρέπει να βρούμε τα σωστά μέσα, ε, μέσα προσαρμοσμένα, αλλά όλα αυτά χωρίς να διακυβεύονται ούτε οι αρχές, η αρχή της ε, μετάθεσης απόσπασης, ούτε της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων και των υπηρεσιών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την εντύπωση ότι μερικές φορές ε, αυτές οι αρχές διακυβεύονται. Για μας η αυτορύθμιση δεν είναι η λύση. Και η πρόταση που συζητείται αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε θα δημιουργήσει ορισμένε δυσκολίε. Όσον αφορά το περιεχόμενο. Ήδη συζητήσαμε τη διάρκεια, δύο χρόνια είπαμε. Προ το παρόν γνωρίζουμε ότι η απόσπαση πρέπει να είναι προσωρινή, το δεχόμαστε. Εφόσον πρόκειται για μια οδηγία του 96 και συζητούμε το θέμα των 24 μηνών. Ένα παράδειγμα για να το εξηγήσω. Γιατί αμφισβητούμε αυτό το γεγονό στη Γαλλία, για παράδειγμα η μέση διάρκεια της απόσπασης είναι 44 ημέρες. Λοιπόν, τι θα αλλάξει με αυτό το όριο. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μακροχρόνια κινητικότητα, μακροχρόνιες αποσπάσεις πέραν των δύο ετών, μέχρι τρία και τέσσερα χρόνια. Αυτό ε, επιτρέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και δεν βλέπουμε ε, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Για... Δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε για τι εταιρείε ούτε για του Γιατί να αλλάξει λοιπόν. επίση επανέρχομαι σε αυτό το θέμα που έλεγε πρωτήτρο συνάδελφο, Υπάρχει εδώ νομικό πρόβλημα αναφορικά με την εφαρμογή του κανονισμού και θα θέλαμε αυτό το θέμα της νομιμότητας να συζητηθεί εις βάθος, διότι προς το παρόν αυτό είναι το πρόβλημα για μας. Όσον αφορά τις αποδοχές, όλοι μας λένε και αυτή είναι η απάντηση που μα δίνεται πάντα, ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι ελάχιστε αποδοχέ. Δεν είναι πρόβλημα. Μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά για ε, όσου αναθεωρούν την οδηγία δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όταν έχετε όμω να εφαρμόσετε τα κείμενα ε, τη πράξη, τότε υπάρχουν τα προβλήματα. Και επιμένω από αυτό, διότι στη Γαλλία έχουμε παρόμοια νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζονται περισσότερα από τι ελάχιστε αμοιβέ και αποδοχέ πέραν δηλαδή της των ελαχίστων αποδοχών. Αυτό ε, στην γαλλική νομοθεσία. Όλοι λένε αν υπάρχει στην γαλλική νομοθεσία μπορεί να υπάρχει και παντού. Και αυτό διότι συζητάμε στα μέλη εταιρείε μας καθημερινά και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εφαρμογή. Διότι όταν οι επιχειρήσεις που ε, στέλνουν αποσπασμένου εργαζόμενου στη Γαλλία και προσπαθούν να καταλάβουν ποια είναι τα ελάχιστα επίπεδα αποδοχών, είναι πολύ δύσκολο να το βρουν ε, για τη μεταλλογική βιομηχανία υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει, αλλά δεν ξέρουν ποια είναι τα σωστά στοιχεία που θα λάβουν υπόψη για να εκτιμήσουν ποια είναι η ελάχιστη αποδοχή. Χρειάζεται χρόνο και σα το λέω διότι το την περμένη εβδομάδα είχα αυτό το πρόβλημα. Η δίκη εργασία την, την περμένη εβδομάδα ζήτησε τη βοήθειά μα. Διότι μα είπε ότι ειλικρινά είναι πολύ δύσκολο να δούμε ποιο είναι το σωστό επίπεδο αποδοχών για του αποσπασμένου εργαζόμενου στον κλάδο μα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολο λοιπόν. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και όταν είσαστε μια εταιρεία 50 ατόμων που στέλνετε ένα αποσπασμένο στο εξωτερικό, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Δηλαδή, πώ να υπολογίζετε το σωστό επίπεδο που προβλέπουν οι συλλογικέ συμβάσει για το ελάχιστο επίπεδο αμοιβών. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και πρέπει να το λάβετε υπόψη όταν αναθεωρείτε την οδηγία. Εν κατακλείδη, πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα τη υπεργολαβία. Ε, είναι ένα πρόβλημα σημαντικό το οποίο παρεμβάλλεται στην αυτονομία μας. Πώς μπορείτε να ζητήσετε σε μια εταιρεία να εφαρμόσετε το αποσπασμένο εργαζόμενο τους όρους που ορίζονται από άλλη εταιρεία που είναι ο βασικός εργολάβος, εργολήτης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος, διότι αλλάζει το πρότυπο ε, που έχουμε ως κοινωνική εταίρη στην Ευρώπη και πρέπει να εξετάσουμε εις βάθος, διότι νομίζω ότι έτσι διακυβεύεται η αυτονομία των κοινωνικών σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Now I would like to ask Mr. Sam Haglund, General, General Secretary, Secretary European... Ευχαριστώ. Ο γραμματέας της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας ε, του κατασκευαστικού τομέα. Όταν υιοθετήθηκε η οδηγία το με την αρχή της χώρας υποδοχής, αυτό δεν ήταν κάτι καινούργιο, γιατί ήδη ξεκίνησε αυτή η αρχή το 1950. Η αρχή της χώρας υποδοχής ήταν βασική για τη δημιουργία της ε, εσωτερικής αγοράς. Αυτή η αρχή εγκαθιδρύθηκε με την ιδέα ότι θα διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός, ότι θα υπάρχει μία ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εταιριών, των ομίλων, των χωρών, όχι όμως βάση της καινοτομίας, αλλά βάση των χαμηλότερων αποδοχών. Αυτά είναι τα επιχειρήματα και πιστεύω ότι οι πατέρες που ίδρυσαν την Ευρώπη είχαν δίκιο. Το ίδιο θα έλεγα και για την οδηγία του 1996. Η οδηγία υποχρεώνει κάποια πράγματα, τα κράτη-μέλη, και τους δίνει και κάποια δικαιώματα. Η υπόθεση Λαβάλ που τελικά οδήγησε στην απόφαση του δικαστηρίου είναι ένα μείγμα αυτών των δύο. Οι ελάχιστες ε, προϋποθέσεις ε, και συνθήκες που θα πρέπει να ισχύουν για όλους, ακόμα και για τους αποσπασμένους και αλλοδαπούς εργαζόμενους και από την άλλη το θέμα των λιγότερο ευνοϊκών συνθήκων που θα μπορούσαν να ισχύουν για τους ε, αποσπασμένους ή αλλοδαπούς εργαζόμενους και είδαμε ποια ήταν η απόφαση ε, στην υπόθεση Λαβάλ. Η επανερμηνία τελικά του άρθρου της συνθήκης που ξαναβλέπει την χώρα προέλευσης και την θέτει αυτή σαν βάση για τις συνθήκες που θα ισχύουν και όχι πλέον την χώρα υποδοχής. Η υπόθεση Λαβάλ είχε και κάποιες άλλες αρνητικές συνέπειες. Η απόφαση που αφορά την Γερμανία και το Λουξεμβούργο, παραδείγματος χάρη. Στις 8 Μαρτίου υπέβαλε η Επιτροπή το σχέδιο πρότασής της και η πρώτη μας αντίδραση ήταν ότι ήταν μια θετική, μια καλή πρόταση αναφέρεται στις ελάχιστες, στις ελάχιστες αποδοχές και βεβαίως αναφέρεται και σε κάποια μοντέλα. Η απόφαση Ρίφερ στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει πλήρως, γιατί τελικά βλέπουμε ότι για 11 χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτό το ελάχιστο μισθό, τις ελάχιστες αποδοχές, η αρχή της χώρας υποδοχής δεν είναι αυτή στην οποία βασίζονται πάντα οι ελάχιστες αποδοχές. Η οδηγία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνεται και να είναι συμβατή με τα διάφορα κοινωνικά μοντέλα των κρατών μελών. Οι τέσσερις χώρες ε, στις οποίες ε, αναφέρεται η υπόθεση Λαβάλ έχουν τελείως διαφορετικούς κανόνες. Το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Γερμανία σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να κάνουν διακρίσεις. Μετά όμως από την υπόθεση Λαβάλ μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Και θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα. Η επικουρικότητα όπως ισχύει στην Δανία. Και έχουν δίκιο εδώ οι Δανείς στις παρατηρήσεις τους. Αναφέρεται στις ελάχιστες συνθήκες και στις ελάχιστες αποδοχές που θα πρέπει να βασίζονται στην εθνική νομοθεσία της χώρας υποδοχής, στην οποία βρίσκεται και εργάζεται ο αποσπασμένο εργαζόμενος. Και δεν νομίζω ότι εδώ μπορούμε να υποψιαστούμε τους δανούς, καθότι στην ιτολογική σκέψη 12 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο ότι το προήμιο και οι ιδεολογικές σκέψεις δεν έχουν την ίδια νομική ισχύ όπως και το κείμενο της ε, νομοθετικής αυτής πρότασης. Οι επιχειρήσεις σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την απόσπαση σαν ένα μόνιμο τρόπο εργασίας με σκοπό να μειωθεί το κόστος του εργαζόμενου. Και τέτοιου είδους ε, ρυθμίσεις, οι οποίες επιτρέπουν αυτές τις αποκλήσεις, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ε, καλές νομοθεσίες. Αν ο σκοπός είναι να μειωθεί το κόστος της εργασίας και να μην τηρηθούν τα δικαιώματα για μια μεγάλη χρονική περίοδο, αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισχύει, ιδιαίτερα αν αυτή η περίοδος είναι τακτική, επαναλαμβανόμενη και ξεπερνάει κάποιο χρονικό διάστημα. Ολοκληρώνω, γιατί έχω μόνο έξι λεπτά. Πρώτον, το θέμα των αποδοχών σε σχέση με αυτή την οδηγία ουσιαστικά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους μόνο τη χώρα υποδοχής και κανένα άλλο ευρωπαϊκό κριτήριο. Δεύτερον, η οδηγία είναι αν θέλετε το ελάχιστο που θα πρέπει να ισχύει και σε κάθε περίπτωση από την πρώτη ημέρα που κάποιος αποσπασμένος εργάζεται σε μια χώρα θα μπορούσε αυτό να τον οδηγήσει στην πλήρη εναρμόνιση με αυτά που ισχύουν για την χώρα αυτή. Θα αναφερθώ επίσης και στην υπόθεση της Φιλανδίας που αναφέρεται στη χώρα υποδοχής και στα ίσα δικαιώματα των αποσπασμένων με τους ε, εργαζόμενους της χώρας υποδοχής. Ευχαριστώ. Πάτρικ Λίμπους από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατών Οικοδόμων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την ανοιχτή συζήτηση για τις αποσπάσεις ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων της οικοδομής Χαίρομαι που λαμβάνω το λόγο στη συνέλευσή σας για να συζητήσουμε για τις επιπτώσεις που έχει αυτό το φαινόμενο στις μικρομεσαίες, για την κινητικότητα και τις αποσπάσεις. Θεωρούμε ότι η αγορά εργασίας της Ένωσης δεν είναι πια η ίδια με το 96. Έχει αλλάξει δραστικά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενσωμάτωση 13 νέων χωρών μελών, με διαφορετικές συνθήκες οικονομικές, κοινωνικές, αμοιβών. Είναι λοιπόν προφανές ότι η επανέναρξη, μάλλον ο επαναπροσδιορισμός των κανόνων επιβάλλεται και ζητάμε γι' αυτό το λόγο την αθεώρηση κανονισμών που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και ίση σημαντικό να επαναπλαισιώσουμε τη συζήτηση για το δικό μας τον κλάδο. Μιλάμε πράγματι για 2 εκατομμύρια εργαζόμενου αποσπασμένου στην Ευρώπη. 44% όμω αυτών των εργαζομένων είναι στην οικοδομή. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα φαινόμενο που αφορά το 5% του πληθυσμού του κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην οικοδομή που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να μην καταστρέψουμε, να μην εξαλείψουμε σύντομα και πλήρως τις θέσεις εργασίας. Το παράδειγμα λοιπόν της οικοδομής στο Βέλγιο είναι εύλοτο. Έχουμε 15.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν τοπικά και έχουμε 15.000 νέους αποσπασμένους τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως μας δείχνουν οι επίσημες στατιστικές της Κομισιόν. Ο τομέας μας χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση στη ζήτηση εργατικού δυναμικού και αφορά βεβαίως την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό βεβαίω έχει επιπτώσεις στους μισθού και των αποσπασμένων αλλά και των ντόπιων εργαζομένων. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να μειώσουμε τις επιπτώσεις και τις κοινωνικές και σε επίπεδο αμοιβών αυτών των φαινομένων ώστε να έχουμε ε, ε, ποιοτικά χέρια ε, ποιοτικέ θέσει εργασία. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με τις ε, επιχειρήσεις που κάνουν αποσπάσεις προσωρινές απλά και μόνο για να μείνουν αγωνιστικές σε επίπεδο τιμών. Σε περίοδο κρίσης, εδώ έχουμε την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στην οικοδομή. Όλα αυτά δυστυχώς δεν μπορούν παρά να συμβάλλουν στην απόρριψη του ευρωπαϊκού εγχειρήματο όσον αφορά την κοινωνία, της κοινωνίας της χώρας μας. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε απώλεια εξειδικευμένων εργατών στις χώρες μας. Έχουμε δηλαδή μόνο ε, εργάτες οι οποίοι εργάζονται τοπικά. Τώρα για τη διάρκεια της απόσπασης θα πρέπει να δούμε ακριβώς τη μέση διάρκεια της απόσπασης στον ε, κλάδο της οικοδομής. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι βρισκόμαστε στις 40 ημέρες. Αυτό αποδεικνύει, θεωρούμε, δύο πράγματα. Μια έλλειψη συνάφειας ή συνέπειας και ότι η πραγματικότητα μας οδηγεί στο να οδηγήσουμε, την, να ορίσουμε μάλλον τη μέγιστη διάρκεια σε συνεργασία με τους εταίρους του κλάδου, ώστε να είναι η διάρκεια αυτή πιο λογική και σε συνεργασία με τις αρχές. Εξάλλου, η ύπαρξη απόσπασης κάτω των έξι μηνών οδηγεί στην παράκαψη αυτών που θα προβλέπει η αναθεώρηση της οδηγίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ενδιάμεση, η προσωρινή εργασία δεν έχει καμία σχέση με, την, με τις αποσπάσεις και ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετά εργαλεία για την παράκαψη της νομοθεσίας μέσω κατάχρησης αυτής της απόσπασης. Χρησιμοποιούνται επιχειρήσεις ενοικίες εργαζομένων για αυτό το σκοπό. Να σας θυμίσω ότι και το Γαλλικό Κοινοβούλιο είχε ένα ψήφισμα που υπέβαλε ο κύριος Σαβαρή όπου έλεγε ότι αυτές οι αποσπάσεις είχαν αυξηθεί θεαματικά 3.000% τα τελευταία χρόνια. Σε σχέση με το επίπεδο των αμοιβών, είναι ξεκάθαρο το ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να αποτελεί το εργαλείο σύγκρισης σε ένα τομέα που παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Διαπιστώσαμε μεγάλες διαφορές σε επίπεδο αμοιβών και πρέπει να δούμε ακριβώ τι γίνεται με τον κοινωνικό διάλογο, με τους κοινωνικούς εταίρους για αυτό το θέμα. Εμείς χαιρόμαστε που υπάρχει ομοφωνία εδώ στην Ευρώπη για την προστασία των εργαζομένων και την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και του αθέμητου ανταγωνισμού. Και μάλιστα από τη στιγμή που σε κάποιες χώρες τα κοινωνικά όρια δεν έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω αυθαιρεσίε. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας και εγώ και η οργάνωσή μα είμαστε στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ όλους για τις ενδιαφέρουσες και επικοδομητικές παρεμβάσεις. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συνεισηγητές. Την κυρία Σαρτιέ και την Άννες Βέριους. Παρακαλώ την κυρία Μωρίν Σαρτιέ να μας μιλήσει. Η έχει ε, δυστυχώς έχεις μόνο δύο λεπτά, Ελιζαπέθ. Ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά, με μεγάλη ευχαρίστηση σας άκουσα τους μεν και τους δε. Και το συμπέρασμά μου είναι ότι τελικά οι εμπειρογνώμονες είναι εξίσου παίκτε όσο και οι πολιτικοί. Θα προσπαθήσω λοιπόν να εκφράσω το πνεύμα της αναθεώρησης αυτής της οδηγίας. Σήμερα η Ευρώπη δεν είναι το Far West. Είναι ένας χώρος όπου πρέπει να οργανώσουμε μια ενιαία αγορά αφενός, αλλά και την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και των πολιτών. Συνεπώς, σε αυτό το πλαίσιο, η αναθεώρηση της οδηγίας έχει κάποιο νόημα προκειμένου να αποφευθούν δύο προσκόμματα, τα οποία αναφέρθηκαν από, τον, από τους μένους τους δε, αλλά είναι δύο εμπόδια, αφενός το κοινωνικό dumping, δηλαδή το να παίζουμε ε, στα μέτρα κοινωνικής προστασίας και τους μισθούς ορισμένων χωρών ή των άλλων χωρών και αφετέρου το να θέμε τον αγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν για να ανταποκριθούν σε πρόσκληση διαγωνισμών τους αποσπασμένους εργαζόμενου οι οποίοι θα αμείβονται με χαμηλότερε αποδοχές, αλλά που μπορούν να ανταποκριθούν και υπόθηκε ε, σε επαγγελματικέ ανάγκες, σε ειδικότητε που δεν υπάρχουν σε ορισμένε χώρες. Υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που λείπουν σε μια χώρα. Ορισμένη ε, εκπαίδευση που λείπει σε μια χώρα ενώ υπάρχει σε μια άλλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει νόημα στο να αναπτύξουμε τις παρεμβάσεις σας και να επικοδομήσουμε από αυτόν. Αναφερθήκατε και σε αρνητικά σημεία, η μεν και η δε. Θα ήθελα όμως όλα αυτά να τοποθετηθούν στο πνεύμα μιας ε, κοινωνικής οικονομίας αγοράς. Η κυρία Κάρτερ από την ΣΕΡΕΣ μας είπε ότι η κοινωνική Ευρώπη χάνει ταχύτητα. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό σήμερα πιστεύω. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να οικοδομήσουμε την κοινωνική Ευρώπη δεν φτιάξαμε, δεν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε την Ευρώπη με βάση την κοινωνική Ευρώπη. Σήμερα όμως υπάρχει ανάγκη αυτής της κοινωνικής Ευρώπης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τη νέα οδηγία. Μέσα σε αυτό το πνεύμα προσπαθούμε να ακούσουμε τους μεν και τους δε και να οικοδομήσουμε πάνω στα όσα μας προτείνεται. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες. Είναι πολύ ενημερωτικό να σας ακούει κανείς και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις σας για να λύσουμε ορισμένα θέματα. Το πρώτο θέμα, το οποίο θεωρώ πολύ ενδιαφέρον, είναι το εξή. και το, στο οποίο αναφέρθηκαν πολλοί παρεμβαίνοντες. Δηλαδή, η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού δεν αφορά μόνο το κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά επειδή υπάρχει έλλειψη ορισμένων ειδικοτήτων. Εάν το δεύτερο ισχύει για την ε, απόσπαση και τη μετακίνηση των εργαζομένων, ποιο είναι το πρόβλημα να έχουν υψηλότερε αποδοχέ αυτοί οι εργαζόμενοι. Εάν ε, ο λόγο αυτής ε, της μετανάστευση των εργαζομένων είναι η έλλειψη ειδικοτήτων, γιατί να μην κερδίσουν περισσότερα. Μπορεί να μην αμείβονται με το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, γιατί να μην μπορούν όμως να μεταναστεύσουν. Το δεύτερο αφορά την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Ορισμένοι ψωμυρογνώμονες αναφέρθηκαν σε αυτό το πρόβλημα. Δεν θα ήθελα να ακούω μόνο προβλήματα. Έχετε και ορισμένε προτάσεις να μας κάνετε. Δηλαδή πώς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε γενικές γραμμές. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσουμε τη φράση που ανέφερε ο κ. Χάκλουγκ, ε, στην αλυσίδα εφοδιασμού. Δεν έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση να κάνετε. Να κάνετε και τέλος ποια είναι η νομική βάση αυτού του πλαισίου. Ένα από τα προβλήματα αυτής της οδηγίας είναι ίσως το εξής. Ενώ αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών ως νομικής βάσης, συνεπώς προστατεύει και τους εργαζόμενους που είναι το αντικείμενο αλλά δεν το αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο το ECG και μήπως θα πρέπει να δώσουμε διτή νομική βάση σε αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον να εκπροσωπεί την ECR που είναι εξάλλου και σκιώδης εισηγήτρια, εκπρόσωπες της ECR δώσω το λόγο στην Μαρτίνα Λαμπάιοβα, άλλη και οδησηγήτρια. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τη Γραμματεία που οργανώνει αυτή τη συνάντηση, εξαιρετικά χρήσιμη για όλους μας. Έχω και ερωτήσεις και σχόλια. Μια ερώτηση προς όλους σας. Έχουμε σήμερα εδώ την ε, πρόταση της Επιτροπής που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Και βεβαίως εδώ έχουμε τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών ε, της Ανατολής, της Ανατολικής Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης και κυρία Λίνακαρ, έχω μία ερώτηση προς εσάς. Μιλήσατε για τις καταχρήσεις, την λανθασμένη εφαρμογή των κανόνων, τις τρευλώσεις στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή η πρόταση θα περιορίσει τις καταχρήσεις αυτές και την κακή εφαρμογή ή αν πρέπει κάτι άλλο να αλλάξει. Συμφωνώ με τον καθηγητή από το Άμστερνταμ που μιλάει για τη διαφάνεια. Διαφάνεια όσον αφορά τις αποδοφιές, παραδείγματος χάρη. Βλέπουμε ότι ο αποσπασμένος εργαζόμενος όταν ενσωματώνεται σε μία αγορά, οι διαφορετικές προϋποθέσεις, όροι και αποδοχές είναι κάτι που αμέσως δημιουργούν το πρόβλημα και συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε. Μιλήσατε επίσης και για το επιπλέον κόστος. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί μιλήσατε για τη φορολογία, το διασυνοριακό κόστος. Πώς το υπολογίζουμε αυτό στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Έχετε κάποια παραδείγματα χωρών. Γιατί από εκεί εξαρτάται βεβαίως το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και η επιπλέον, το επιπλέον κόστος που οφείλεται στη φορολογία βεβαίως εδώ οδηγεί σε κάποιες επιλογές. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Ευχαριστώ Μαρτίνα. Ειρήνια Ρόνια Κάρης είναι επίσης και όδηση εισηγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ σε όλους όσους είναι σήμερα εδώ όλους τους εμπειρογνώμονες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να ακούσει όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις και έχω δύο πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα να σας κάνω. Πρώτον, απευθύνομαι σε όλους τους εμπειρογνώμονες. Η απόσπαση εργαζομένων είναι ένα φαινόμενο περιορισμένο στο χρόνο. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Οι πολιτικοί συνήθω λένε ότι πρόκειται για ένα μέσο πρόθεσμο φαινόμενο. Εσείς λέτε ότι δεν είναι καλή η πρόταση της Επιτροπής. Πώς όμως μπορούμε να περιορίσουμε αυτές τις αποσπάσεις έτσι ώστε όντως να είναι περιορισμένες στη διάρκεια. Θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα δηλαδή της διάρκειας αυτής της απόσπασης. Ποια είναι η καλή κατά την άποψή σας διάρκεια. Και για την Business Europe έχω μία ερώτηση. Αναθεώρηση της οδηγίας κάνουμε εδώ. Και η ερώτησή μου είναι εξή: Οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας, γιατί μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι οι επιχειρήσεις είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους και με τους εργαζόμενους επιτόπου οι επιχειρήσεις συνήθως υπόκεινται στις συλλογικές συμβάσεις, εκτός εάν δεν έχουν την έδρα τους στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέκα. Δεν είναι εδώ η συγγήτρια. Ζητώ συγγνώμη. Για μας υπάρχουν διάφορες ανησυχίες που θα πρέπει να απαντηθούν για να είναι αποτελεσματική αυτή η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Και μία από τις ερωτήσεις που θέλω να κάνω στην κυρία Χόκ είναι το θέμα του κενού που συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την οδηγία. Δηλαδή τα άτομα τα οποία για κάποιες συμβάσεις μπορούν να φύγουν από τη χώρα τους και να πάνε σε μια άλλη χώρα και να εργαστούν εκεί. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις περιπτώσεις αυτές, να θέσουμε όρια και να μειώσουμε και το φάσμα ισχύω αυτών των συμβάσεων. Και η ερώτησή μου είναι, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποια άλλα στοιχεία σε αυτή την πρόταση είτε να εξειδικεύσουμε κάποιους τομείς. Ευχαριστώ. Λαουρά Τζιά. Και αυτή είναι η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε και πάλι ένα θέμα το οποίο έχει αφήσει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Και ακούγοντα τις διάφορες απόψεις των εκπροσώπων συμφερόντων και πανεπιστημίων είναι σαφές ότι υπάρχει μια βασική δυσκολία εδώ. Εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο την κυρία Μπόη, θυμάμαι το όνομά της, καλά, που ανέφερε το θέμα των αμοιβών και μίλησε για αυτή την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ κρατών και κοινωνίας πολιτών. Πώς εμείς θα μπορούσαμε να υποβάλουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για να ξεπεράσουμε αυτό το διέξοδο. Γιατί συμφωνώ με αυτό που είπε η Μαρτίνα προηγουμένω. Το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο για να βρούμε μια κοινή θέση. Να πω κάτι επίσης σε σχέση με τη διετία. Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων από το νομέα της οικοδομής μας έλεγαν για μία περίοδο απόσπασης 40 ημερών. Εδώ λοιπόν πώς θέλουμε να το λύσουμε αυτό από τη στιγμή που μιλάμε για επέκταση της απόσπασης μέχρι 24 μήνες, δύο έτη. Και αυτά που λέει η κυρία Γιουγκέριους επίσης τα συμμερίζομαι, γιατί νομίζω ότι πραγματικά έθιξε τα τρία πιο κρίσιμα ζητήματα. Επειδή εδώ λοιπόν έχουμε και πανεπιστημιακούς αλλά και εκπροσώπους ε, συμφερόντων, θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς θα μπορούσαμε να καλύψουμε αυτά τα κενά που δημιουργούν αυτές τις ρογμές. Η προηγούμενη οδηγία είχε διαφορετική θεματολογία Αν θέλουμε λοιπόν να καλύψουμε τα ενδεχόμενα κοινά με την τωρινή αναθεώρηση, τότε θα πρέπει οι χώρες μέλη περισσότερο να ασχοληθούν με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας παρά με τις αλλαγές από τις οποίες θα προσδοκούσαν. Ευχαριστώ. Ντομινίκ Μαρτίν τώρα από το ΓΕΝΕΦ. Είναι και σκιώδης συζητητή μας επίσης, ο κ. Μαρτίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση ήρθαν προσωπικότητες που μας παρουσίασαν τις ερευνές τους, αλλά εγώ διακρίνω κάποια κακοφωνία. Οι μεγάλοι εργοδότες είναι αντίθετοι, όπως καταλαβαίνουμε. Και οι μικρομεσαίες του PTP είναι υπέρ, γιατί αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης. Βλέπουμε επίσης και ότι οι ερευνητές δεν συμφωνούν μεταξύ του. Ένας μάλιστα μας είπε ότι οι αποσπασμένοι είναι πιο ακριβοί για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Αυτό θα πρέπει να το αποδείξετε, έτσι. Διαφορετικά θα πρέπει να σταματήσει αύριο το φαινόμενο των αποσπασμένων. Η κυρία Σαρτιέ. Ε, το προηγουμένως ότι η Ευρώπη δεν είναι αγραία δύση. Ναι, βεβαίω. Νοέμβρη λοιπόν καταλάβατε το 2016 Νοέμβριο ότι η Ευρώπη είναι αγριαδίση, είναι κοινωνικό ντάμπι και είναι η Ευρώπη που εσείς ήδη χτίσατε. Α, και μετά τι γίνεται. Α, για κοίτα. Καταλάβαμε ότι ξέχασαμε να φτιάξουμε την κοινωνική Ευρώπη. Εσείς θέλατε να μεγαλουργήσετε με την Ευρώπη των 10, των 12, των τώρα 27, 28 Κυρία Μωράσου όμως είναι κρίμα που χρειάστηκαν 30 χρόνια να το καταλάβετε. Ντομινίκ, λέει πρόεδρος Ντομινίκ, σε παρακαλώ μπορείς να ολοκληρώσεις. Ναι, κάνω διαπίστωση, δεν έχω ερώτηση, έκανα μια διαπίστωση εδώ. Και βρίσκω ότι οι δύο συνεισηγητές είναι πολύ αξιόλογοι και πολύ θαραλέοι. θα δείτε ότι σε λίγο όρος και έτε και εμείς. Γιατί στην ουσία δεν θα γίνει τίποτα. Θα συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να απασχολούν τους και να μετακινούν τους εργαζόμενους αυτούς και τελικά ακούσαμε και προηγουμένως εδώ ότι στις μικρομεσαίες έχουν καλύτερα αποτελέσματα και γι' αυτό θα σταματήσει το φαινόμενο. Έχουν περισσότερα κέρδη με τι αποσπάσει. Και ότι στην ουσία αυτό που ε, εδώ είναι ακριβώ οι αμοιβέ των, εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα... Τώρα δίνω το λόγο στα μέλη. Δυστυχώ έχετε μόνο ένα λεπτό. Και παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το χρόνο σα, επειδή δεν έχουμε πλέον χρόνο. Πρώτα απ' όλα, Παλάμα Λοπέ Μπεμέιο. Ε, Πρόεδρε, Το πρόβλημα της τωρινής οδηγίας δεν είναι η, η μη εφαρμογή. Είναι το ότι έχει μετατραπεί σε εργαλείο κοινωνικού ντάμπινγκ στις χώρες μέλη. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν καν μεταφέρθηκε η οδηγία σε διάφορες χώρες. Οπότε να δούμε τι γίνεται στις οδικές ας πούμε μεταφορές όπου η Ένωση αντιτάχθηκε στην καταβολή κατώτατου μισθού σε Γαλλία-Γερμανία με τις αποσπάσεις βλέπουμε ότι στην ουσία έχουμε να κάνουμε μια δία κατανακαστική μετανάστευση εργαζομένων που είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν σε τρίτες χώρες σε χειρότερες συνθήκες εργασίας. Και θα δείτε ότι λόγω κρίσης οι αριθμοί είναι Ευχαριστώ λοιπόν το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για τη βόλησή του να προωθήσουν αυτή την πρόταση αναθεώρηση τη οδηγία, που περιλαμβάνει θετικέ αρχές όπως το δικαίωμα για την ίδια αμοιβή και την ε, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων. Ναι, Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Υπάρχουν όμω πτυχέ που θα πρέπει να διορθωθούν. όπω ο μέγιστο χρόνο απόσπαση ή η συλλογική συμβάση. Ευχαριστώ. Κατόπιν, Χέζος Νίλσον. Eftersom Marita Ulvskog inte kunde vara här så tar jag tillfället i akt att säga några ord som svensk socialdemokrat. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Είμαστε σε γενικέ γραμμέ ικανοποιημένοι με τι προτάσει που έγιναν. Μιλάμε για τις αποδοχές, αλλά υπάρχει ο κίνδυνο η κάθε χώρα να ερμηνεύσει αυτές τις προτάσεις ανάλογα με το τι ισχύει στην ε, κάθε χώρα. Και όλα τα κράτη-μέλη δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ενιαία ερμηνεία. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να φτάσουμε σε μια καθολική ερμηνεία. Σκεφτείτε παραδείγματο χάρη ότι σήμερα στι χώρε ισχύουν οι συλλογικέ συμβάσει και ότι υπάρχουν εκατοντάδε κλάδοι για εκατοντάδε διαφορετικέ ρυθμίσει και ε, συλλογικέ διαπραγματεύσει που οδηγούν σε, κάποιες, ε, σε κάποια αποτελέσματα που ισχύουν όμω σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν θα διασφαλίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα, τα βασικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην απεργία, παραδείγματο χάρη και οι ελάχιστε αποδοχέ. Αυτά είναι κατά των βασικών αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, ομιλητές. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, θα ξεπεράσουμε το θέμα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε κοινέ ε, συλλογικές συμβάσεις που αφορούν τη μισθοδοσία και τις αποδοχές και τα δικαιώματα. Αυτά αριθμίζονται με τρόπο εθνικό, κλαδικό, ανάλογα με τον τομέα της εταιρείας. Υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά μεγάλες διαφορές και στο επίπεδο αλλά και στην, στο σύστημα εκπροσώπησης παραδείγματος χάρη. Από τη μία χώρα στην άλλη διαφέρουν πάρα πολύ τα συστήματα εκπροσώπησης. Κυρία Βαν Κόκ, έχω μία ερώτηση. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι η αρχή ίση αποδοχή δεν εγκρίνεται κατά την άποψή σας δεν ε, είναι εγγυημένο στην πρόταση της Επιτροπής. Τι θα προτείνατε για να υπάρχουν κάποιες εγγύησεις. give the floor, ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μα είπαν ότι δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία επειδή όλα ήταν θέμα εφαρμογής αλλά τουλάχιστον τρία σημεία πρέπει να αναθεωρηθούν από νομική άποψη. Πρώτα απ' όλα, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις εταιρείε χρηματοκιβώτια, που είναι μεγάλο κακό, η σχέση δηλαδή, σημαντική σχέση μεταξύ του μισθωτού και του εργοδότη. Δηλαδή να υπάρχει μια αρχαιότητα τουλάχιστον τριών μηνών για να καταπολεμήσουμε αυτές τις εταιρείε γραμματοκιβώτια, αλλά να εξασφαλίσουμε και την ποιότητα των εργαζομένων ε, της δουλειάς. Δεύτερον, για να καταπολεμήσουμε πράγμα, αυτές τις τρεις γραμματοκιβώτια είναι το θέμα του κύκλου εργασιών «Αναχώρα» δεν θα πρέπει να εισαχθεί μία αναφορά προκειμένου οι εταιρείε που στέλνουν αποσπασμένους να έχουν τουλάχιστον 25% ε, κύκλο εργασιών σε μία δεδομένη χώρα για να μην πάλι πέσουμε στην περίπτωση εταιρεών που κάνουν το γύρο των χωρών και κάποια μέρα εξαφανίζονται και δεν βρίσκουμε τις κοινωνικές τους παροχές. Τρίτο σημείο, θα πρέπει να διευθυνθεί το θέμα των αποδοχών και στο κείμενο δεν είναι ακόμα σαφές σήμερα. Επειδή εάν υπόθηκε προηγουμένω ότι οι επιχειρήσει αποστολή πληρώνουν για τη στέγαση ε, και την αισθήση κτλ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι επιχειρήσει υποδοχή θα πρέπει να πληρώνουν. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει, επειδή τα πράγματα δεν είναι σαφή, αυτό προστίθεται ή αφαιρείται από την αμοιβή του εργαζόμενου. Ενώ αυτό θα πρέπει να ξεχωριστεί, ε, θα πρέπει να προσθεθεί στην αμοιβή. Αυτό όμω δεν είναι σαφέ το κείμενο. Γι' αυτό στο έγγραφο τη Επιτροπή πρέπει να είναι απόλυτα σαφέ να πούμε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 να ρωτήσω το εξή. Συμφωνούμε μεταξύ μα ότι αυτό το θέμα, αυτή η προβληματική δεν έχει να κάνει μόνο με Ανατολική ή Δυτική Ευρώπη. Βλέπουμε ότι πολλές αποσπάσεις, ε, ίσως περισσότερες ε, αφορούν την Πολωνία, αλλά δεύτερη είναι η δυτικη ευρωπη βλεπουμε οτι πολλέ αποσπάσει ε ισως περισσοτερες Μετά, τι γίνεται με τις ε, συνθήκε ίση αμοιβή. Πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό πώ θα μπορούσαμε να το πετύχουμε σε εθνικό επίπεδο μάλιστα και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό. Οπότε έχουμε αυτό το φαινόμενο με διαφορά στην αμοιβή. Εγώ ίδιος έχω συνεργάτες και βοηθούς οι οποίοι αμείβονται διαφορετικά εδώ στις Βρυξέλλες και στην χώρα μου την ε, Ουγγαρία ας πούμε. Τώρα, το πρόβλημα με την οδηγία αυτή είναι το πώς εφαρμόζεται και πώς σχετίζεται με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Νομίζω αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Τελευταία ερώτηση. Κοινωνικό dumping και αθέμητος ανταγωνισμός. Τι σχέση έχουν αντίστοιχα με την οδηγία για τους αποσπασμένους, γιατί εγώ εδώ φοβάμαι ότι μπερδεύουμε τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά νομίζω ότι δεν αφορούν άμεσα την οδηγία αυτή για τους αποσπασμένους. Μετά για τις ε, επιχειρήσεις αυτές που είναι γραμματοκιβώτια. Θα ήθελα εδώ να ακούσουμε και προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για την συμβολή τους. Να πω ότι διαφωνώ με την πρόταση αυτή. Χαρακτηρισμό της πρότασης αυτής ως εφιάλτη. Νομίζω ότι πάμε πια σε συνθήκες εργασίας Δεκάτου του αιώνα όταν προσπαθούσαμε να καταργήσουμε την παιδική εργασία. Πρέπει να ενημερωθεί, να επικαιροποιηθεί αυτή η οδηγία, ιδιαίτερα όσον αφορά την φύση της απόσπασης, αλλά και στο θέμα των αμοιβών. Να ρωτήσω λοιπόν, γιατί, για ποιο λόγο ένας Ολλανδός έχει επίδομα για βαρέα και ανθυγίνα, νυχτερινή εργασία κτλ. Γιατί δεν ισχύει, ας πούμε, και για κάποιε μητέρε οι οποίε εργάζονται στον ίδιο χώρο εργασία, που δουλεύουν υπό τι ίδιε συνθήκες εργασία. Πρώτη μου ερώτηση αυτό προ του ηγητές. Και δεύτερον, ανεξάρτητα με του κανόνε στου οποίου θα καταλήξουμε, με απασχολεί και το θέμα τη εφαρμογή των κανόνων στου οποίου θα καταλήξουμε. Θα ήθελα λοιπόν οι ηγητές να μα πούν τη γνώμη του για το πώς οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας θα μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστά τους κανόνες που θα συγκροτήσουμε. Αυτά που θα κάνουμε θα μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστά στην πράξη. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες μας. Έχετε τέσσερα λεπτά ο καθένας από εσά για να απαντήσετε στα ερωτήματα ναι, με την ίδια σειρά. Uh, Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τις ερωτήσεις που μας κάνετε. Δεν έχω βέβαια το χρόνο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη σειρά με την οποία τέθηκαν οι ερωτήσεις. Συμφωνώ με την κυρία Αγγέριος. Φυσικά και η μετανάστευση πολλές φορές είναι το αποτέλεσμα έλλειψης κάποιων δεξιοτήτων και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους αποσπασμένους για να καλύπτουμε αυτά τα κενά δεξιότητες, δηλαδή που δεν υπάρχουν στην τοπική αγορά. Το θέμα της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων. Αυτό το βλέπουμε ήδη Κάποιες μόνο συλλογικέ συμβάσεις είναι δεσμευτικές για τον φορέα παροχής ε, υπηρεσιών, ιδιαίτερα για την περίπτωση αποσπασμένων και τους εργαζόμενους στη χώρα στην οποία εργάζονται. Αυτό ισχύει για τις αποδοχές, για το ωράριο εργασίας, για τις συνθήκες εργασίας νομική βάση. Βέβαια πρέπει να διευρυνθεί έτσι ώστε όταν προκύψει ένα νέο θέμα, όταν υπάρχει μια νέα προσφυγή στο δικαστήριο, να μπορούν να ληφθούν υπόψη, όπως ακριβώς έγινε και με την παροχή υπηρεσιών, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Να υπάρχουν οι ίδιες ευθύνες Ποια είναι η καλύτερη λύση, μας κάνατε αυτή την ερώτηση, νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια ακρόαση που θα ξεπεράσει κατά πολύ τις δύο ώρες, είναι πολύ ευρύ το θέμα και δεν πρόκειται να το θίξω καθόλου. Αναθεώρηση, θα απαντήσω ότι εξαρτάται σε τι θα καταλήξουμε τελικά σε αυτήν την μεταρρύθμιση αναθεώρηση, γιατί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα όπως το dumping, αλλά δεν το κάνουμε για άλλα θέματα όπως τη μερική απασχόληση και το θέμα του dumping. Με κάθε σεβασμό προς τα μέλη του Κοινοβουλίου που έθιξαν το θέμα αυτό, θα πω ότι και εμείς θεωρούμε ότι πρώτα πρέπει να διορθώσουμε την οδηγία και μετά να αρχίσουμε να κοιτάμε πώς εφαρμόζεται. Το θέμα της διαφάνειας βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τα θέματα της ε, εφαρμογής του κατά πόσο είναι δεσμευτική αυτή η οδηγία, όμως έχουμε σε πολλά κρατημέλη στοιχεία και πληροφορίες που θα πρέπει να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον πιο αποτελεσματικό. Πολλά από αυτά που άκουσα ήταν σχόλια. Δεν ξέρω ποιος είπε ότι δεν είναι θέμα Ανατολής Δύσης. Ναι, βέβαια. Η Ανατολική και η Δυτική Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσουν μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και βλέπουμε ότι για κάποιο λόγο οι εταιρείες των νέων κρατών μελών της Ανατολικής Ευρώπης είναι λίγο πιο ικανή στο να παρεκκλίνουν των κανόνων. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, εκπροσωπώντας τις ε, εταιρείε ε, νομικής μορφής, ε, τις εταιρείε απόσπασης εργαζομένων κτλ. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποσπαστεί παράνομα. Οτιδήποτε κάνουμε για να τους καταπολεμήσουμε είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι πολλά από τα θέματα που θίξατε συζητήθηκαν σε σχέση με την ε, οδηγία εφαρμογής. Υπάρχει αυτή η οδηγία εφαρμογής και διαπιστώνουμε ότι δεν υλοποιείται, διότι η σημασία δίνεται τώρα στην αναθεώρηση τη οδηγία. Αυτό προσπάθησα να σα εξηγήσω. Και γι' αυτό στράφηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντα του να μα υποστηρίξει προκειμένου αυτή η οδηγία εφαρμογή να είναι λειτουργική. Διότι πρέπει να λειτουργήσει. Τώρα, για το θέμα των αποσπασμένων εργαζόμενων. Αυτό είναι ένα γεγονό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μας βοηθάει στο να καταπολεμήσουμε τις παράνομες εταιρείε ή τους παράνομους αποσπασθέντες. Αυτό είναι το πρόβλημα για μας. Δημιουργεί προβλήματα για τις, ε, ε τις εταιρείε που λειτουργούν ένομα με νόμιμους αποσπασμένους. Προσπάθησα να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Γνωρίζουμε ότι η απόσπαση υπάρχει και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, αλλά ως επιχειρήσεις προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα, για την κοινωνική ασφάλιση που αναφέρθηκε από άλλου προλαλήσαντε, και εγώ προέρχομαι από τη Δανία και πρέπει να ομολογήσω σε αυτήν την αίθουσα ότι αντιπροσωπεύω μια χώρα που είναι ο ε, το, που χάνει το μεγαλύτερο κοινωνικό dumping στην Ευρώπη. Αλλά η αλήθεια σε όσα υπόθηκαν είναι ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα ε, στην οδηγία των αποσπασμένων εργαζομένων και στους κανονισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Αλλά δεν έχουμε πρόταση από την Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλιση. Γι' αυτό σας κάνω έκκληση. Παρακαλώ να δούμε τι προτείνει η Επιτροπή. Και μετά ίσως βρεθούν λύσεις που θα διασυνδέουν την απόσπαση και την κοινωνική ασφάλιση. Ίσως εκεί βρεθεί η λύση. Οπωσδήποτε θα εξετάσουμε αυτό το θέμα αλλά μας χρειάζεται η πρόταση της Επιτροπής και για την κοινωνική ασφάλιση. Νομίζω παράσεις εδώ αναφέρθηκε σε πολλά παραδείγματα. Πολλά είχαν συζητηθεί σε σχέση με την οδηγία εφαρμογής και αυτό πάλι είναι κατά πόσον ε, αφορά την απόσπαση, την οδηγία απόσπαση, με συγχωρείτε. Δεν θα πω αν είναι η καλύτερη λύση, αλλά αυτή ήταν η πολιτική απόφαση. Σας παρακαλώ λοιπόν να έχετε υπόψη ότι αυτό που θέλουν οι εταιρείε είναι νομική σαφήνεια. Να ξέρουν ποιοι είναι οι κανόνες που εφαρμόζονται. Το να αλλάζει κανείς συνέχεια τους κανόνες και λυπούμε ότι, το επαναλαμβάνω συνέχεια, είναι εφιάλτης για τις εταιρείε. Το είπα και πρωτήτερα. Αυτό σε σχέση με την αλλαγή της σύμβασης συνέχεια, των συμβάσεων συνέχεια. Αυτό είναι ένας μεγάλος εφιάλτης για τις εταιρείε και τους υπαλλήλους. Ε, είναι δύσκολο για μας και για έναν Δανό που πάει στη Γαλλία αλλά και για έναν Γάλλο που πάει στη Δανία το γεγονός ότι δεν ξέρει τι ισχύει κάθε φορά αυτό είναι δύσκολο. Η Ευρώπη είναι περίπλοκη. Έχουμε την οδηγία πρέπει να τη βελτιώσουμε. Ε, εξ ονόματος του Business Europe, θέλω να σας πω ότι είμαστε ανοιχτοί και διαδεθειμένοι να εξετάσουμε την πρόταση της Επιτροπής, η οποία όμως θα πρέπει να μας δώσει και ορισμένες προτάσεις για την κοινωνική ασφάλιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Άκη Φων καθηγήτρια, έχει το λόγο. Λέγομαι Άκη Είμαι από το βόρειο τμήμα της Ολλανδίας, από μια μειοψηφική κοινότητα και μειοψηφική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προφέρετε το όνομά μου, ακόμα και για, τις, για τους Ολλανδούς. Το θέμα του equal pay των ίσων αποδοχών και γιατί αυτό δεν προστατεύεται από την πρόταση της Επιτροπής. Θα σας εξηγήσω. Οι εγγυήσει θα πρέπει να δίνονται από τις συλλογικές συμβάσεις και από την νομοθεσία και αυτό καλύπτεται για ένα συγκεκριμένο τομέα. Σε πολλές χώρες αυτό δυστυχώς δεν ισχύει πλέον. Σε κάποιες δεν υπάρχει και σε κάποιες δεν ισχύει πλέον λόγω της κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Οι συλλογικές συμβάσεις σήμερα έχουν ε, αντικατασταθεί από άλλου είδους συμβάσεις και διευθετήσεις και συμφωνίες. Το θέμα λοιπόν του καθορισμού των αποδοχών που ήταν αν θέλετε αρχικά το μέλημα του μονομοθέτη, δηλαδή να γίνουν σεβαστές οι εθνικές παραδόσεις, συνήθειες και νομοθεσία. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθούν σήμερα σαν περιορισμοί διότι η ιδέα ήταν να συμπεριληφθούν ακόμα και αυτές οι διαφορετικές σχέσεις ε, και συμβάσεις εργασίας, όπως παραδείγματος χάρη όταν ε, παρεμβαίνει ένας ε, υπεργολάβος ή ένας εξωτερικός φορέας. Το θέμα των αποσπασμένων εργαζόμενων βεβαίως πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τις εθνικές παραδόσεις, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα της αγοράς, την ε, ύπαρξη ημί φορέων ε, εξωτερικής ανάθεσης, είτε ε, υπεργολα... σχέσεις υπεργολαβίας. Και σίγουρα θα πρέπει να βρεθούν λύσεις αποτελεσματικές, πιο αποτελεσματικές από αυτή που προτείνεται εδώ και που σχεδιάζεται εδώ, διότι η σημερινή πρόταση Επιτροπής ουσιαστικά προσκρούει σε όλες τις εθνικές παραδόσεις και νομοθεσίες. Υπάρχουν λοιπόν πολλές τέτοιες περιπτώσεις αποσπάσεων. Το στέλεχος το πολύ καλοπληρωμένο που στέλνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες, ένας εργαζόμενος από την Ευρώπη που θα πάει με μια ευρωπαϊκή σύμβαση να εργαστεί στην Αφρική. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει αυτό που θα ισχύει να ισχύει παγκοσμίω και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα τώρα της απόσπασης και των δεσμευτικών ε, προϋποθέσεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ισχύει για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Καταρχήν άπτεται της ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να μην αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα. Αλλιώς θα αρχίσουν να αλλάζουν τα πάντα, ακόμα και το ωράριο εργασίας, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί, παραδείγματος χάρη, στην επιθυμία ενό εργαζόμενου να παραμείνει με την οικογένειά του. Το θέμα είναι τι προστασίες θέλουμε για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε απόσπαση και άσχετα με το τι ισχύει ε, στην μία την άλλη χώρα. Και αυτό μπορεί να γίνει στο άρθρο 1 και κατόπιν μπορούμε να συζητήσουμε για τον περιορισμό της διετία κτλ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να θέσουμε εδώ σε αμφισβήτηση ένα σύστημα το οποίο έχει πολύ πιο ευρύ αποδοχή και ισχύ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Μπενιό, ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω τα ερωτήματα που μου απευθύνατε πρώτα σε μένα και μετά να σχολιάσετε τα υπόλοιπα. ρωτήσατε πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί Δεν θα έχουμε αυτό συμπληρωματικό κόστος. Νομίζω μία πιθανή απάντηση έδωσε η κυρία Κέριους που έλεγε ότι οι περισσότερες αποσπάσεις οφείλονται στην έλλειψη αυτών των προσόντων στις χώρες υποδοχής. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τοπικός ανταγωνισμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο νόμος είναι διαφορετικός. Αν υπήρχε ανταγωνισμός ντόπιο, τότε η χώρα θα, συγγνώμη, επιχείρηση θα έπρεπε να πληρώνει κάποια επιδόματα που τώρα η Κομισιόν θέλει να περιλάβει στις αμοιβέ. Οπότε προτιμούν να πληρώσουν αυτό το συμπληρωματικό κόστος από ότι αυτά τα επιδόματα επιχείρηση. Και η κυρία Γκλαμπάγιοβα αυτό που ρώτησε ασχολείται στο εξή. Να δώσω δύο παραδείγματα. Υπάρχει μια διαφορά στους κανόνες που ισχύουν τοπικά, που αφορούν τις τοπικές επιχειρήσεις και υπάρχουν και κάποιες δαπάνες που αφορούν μόνο τους αποσπασμένους και το οποίο εγώ θεωρώ ως φραγμό για την παροχή υπηρεσιών. Ας πούμε στη Γαλλία υπάρχει μια επιβάρυνση που αφορά συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό αφορά Ξένου εργαζόμενου, αλλά και Γάλλου. Υπάρχει όμως επίσης και μια επιβάρυνση όσον αφορά την κοινοποίηση που θεσπίστηκε πρόσφατα 50 ευρώ αναποσπασμένο. Αυτά είναι λοιπόν τα χρήματα που η τοπική επιχείρηση δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ποτέ και που μια ξένη επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει. Αυτό θεωρώ εγώ ως φραγμό για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Και μιας και μιλάμε για φραγμούς, να πω και κάτι σχετικά με αυτά που ο κύριος Μπάλας, ο οποίος προτείνει κάτι νέο που δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει ένας ελάχιστος κύκλος εργασιών στην χώρα προέλευσης όσον αφορά τους εργαζόμενους, αν κατάλαβα καλά. Αυτή η ιδέα προέρχεται νομίζω από το συντονισμό κοινωνικής ασφάλισης. Άλλη μια ιδέα, το 24μενο, αφορά και προέρχεται και αυτή από τον συντονισμό των κοινωνικών ασφαλίσεων. Εγώ όμως το εκλαμβάνω σε εξή ότι ανεξάρτητα από τη χώρα μέλος στην οποία έρχεται την εργασία σας ή την επιχείρησή σας, εσείς θα πρέπει να είστε σε θέση να παράσχετε υπηρεσίες σε άλλες χώρες μέλη. Εύκολα λοιπόν, μέχρι τη θέσπιση αυτού του κανόνα, θα έχουμε πολύ κινητικές ή ευκίνητες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα έχουν 20% κύκλο εργασιών στις χώρες που παρέχουν υπηρεσίες, επειδή είναι πολύ ευκίνητες. Εγώ δεν θα ήμουν και τόσο υπέρ αυτών των όριων. Όρια που είναι και αυτά από μόνο τους φραγμοί. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Και μια τελευταία παρατήρηση, μια και έχω μόνο 10 δευτερόλεπτα. Δεν ήταν δική μου μόνο η έρευνα. Όταν η Κομισιόν επέβαλε αυτή την πρόταση, υπήρχε ένα κενό δεδομένων. Όχι μόνο στη δική μου έρευνα, αλλά είχαμε και μια πρόσφατη του Ιούνιου του 2016 Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας της Γαλλίας, όπου κατέδειξε ότι ο Γάλλος απασχολούμενος είναι πιο ακριβώς, διορθώνει ο μιλητής, είναι λιγότερο ακριβώς από έναν Πολωνό αποσπασμένο. Το ίδιο ισχύει φαντάζομαι και το κόστος εργαζομένων από Πορτογαλία, Ισπανία. Διακόπτη η πρόεδρο. Παρακαλώ τελειώστε. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ, λέει ο μιλητή. Α, ναι. Τελευταίο. Ψάξτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία. Γιατί νομίζω απλά και μόνο εδώ μαντεύουμε. Είμαστε μάντις. Πολλά θέματα θίξατε και πολύ ενδιαφέροντα. Είναι κρίμα που δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, αρκετά γεγονότα. Εάν μπορείτε, αφού ζητήσετε στους εμπειρογνώμονες, να στείλετε στη γραμματεία και την παρουσίασή σας και τα ερωτήματά σας, θα, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτού του πολύ περίπλοκου θέματος. Στρέφομαι τώρα στην κυρία Δελφίνου Ρουντέλη. Ευχαριστώ. Ορισμένε παρατηρήσει. Θα ήθελα να επανέλθω στο γεγονό ότι είναι λίγο δύσκολο για κάποιους σαν και εμένα όταν μιλάτε για απόσπαση. Κατευθείαν οι υπόλοιποι μιλάνε για κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό είναι δύσκολο για μας και κουραστικό. Διότι όταν συζητάτε με τις εταιρείε μέλη, όπως κάνουμε εμείς καθημερινά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν κάνουν απόσπαση εργαζομένων, δεν λαμβάνουν εργαζομένους, για... όχι επειδή κάνουν κοινωνικό ντάμπινγκ και για πολλούς άλλους λόγους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε αυτούς που στέλνουν ε, αποσπασμένους εργαζόμενους με νόμιμο τρόπο. Και θα ήθελα να απαντήσω σε ένα σχόλιο. Είναι εύκολο να αντιπαραθέτει κανεί τι μεγάλε και τι μικρέ εταιρείε. Στο δικό μου τομέα, οι περισσότερε από 85% είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και αυτέ οι εταιρείε στέλνουν ε, αποσπασμένου εργαζόμενου. Η απόσπαση δεν είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από ορισμένου, από του μεγάλου μόνον. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Και πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφεί από αυτού. Διότι μερικέ φορέ έχω την εντύπωση ότι τα έχουμε ανακατέψει όλα μαζί αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι η απόσπαση πρέπει να συνδέεται πάντοτε με την παράνομη εργασία και με το κοινωνικό ντάμπινγκ. Βεβαίω, σε ορισμένε περιπτώσει, οι οποίε είναι φοβερέ, τι αναφέραμε, ε, υπάρχει αυτό και εδώ πρέπει να βρούμε λύσει. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση, το παραλαμβάνω, δεν θα μα βοηθήσει να βρούμε τη σωστή λύση. Αναφέρθηκα σε αυτή την οδηγία εφαρμογή οι συνάδελφος από το Business Europe αναφέρθηκε στην κοινωνική ασφάλιση και στους κανονισμούς. Νομίζω ότι αυτό είναι ο κανονισμός κοινωνικής ασφάλισης είναι το σωστό εργαλείο που μπορεί να μας δώσει μια λύση και δυστυχώς η Επιτροπή δεν παρουσιάζει αυτή την, ε, την οδηγία του 96 με τον κανονισμό για την κοινωνική ασφάλιση. Οτιδήποτε προκύψει από τη συζήτηση εδώ πρέπει ένα να έχουμε υπόψη οτιδήποτε αποφασιστεί θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμο. Γιατί τελικά. Γιατί ορισμένες φορές η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται. Επειδή δεν είναι εφαρμοστέα. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Αν πάρετε τη διάταξη για την υπεργολαβία, για να είμαστε δίκαιοι, εάν διαβάσετε το σχετικό άρθρο, χρειάζεται χρόνο για να καταλάβετε τι σημαίνει. Και όταν έχετε τέτοιου είδους διατάξεις σε ένα νομικό κείμενο, αυτό δεν είναι παραδεκτό, διότι τελικά, εάν μία επιχείρηση πρέπει να στραφεί σε ένα νομικό εμπειρογνώμο για να καταλάβει αν θα εφαρμόσει ή όχι αυτή τη διάταξη, αυτό δεν λειτουργεί. Πρέπει να είναι οι διατάξεις απλές. Πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη εύκολα. Νομίζω ότι ένας ευρωβουλευτής έθιξε αυτό το θέμα. Δηλαδή η οδηγία εφαρμογής μπορεί εύκολα να ειναι οι διαταξει απλες πρεπει να μπορουν να εφαρμοστουν στην πραξη ευκολα νομιζω οτι ενας ευρωβουλευτή εθιξε αυτο το θεμα δηλαδη η οδηγια εφαρμογή μπορει ευκολα να γινει κατανοητη απο του επιθεωρητέ εργασία με τα χαρά να το συζητήσουμε μετά από τι συνεδρίε. Έχω πολλά παραδείγματα. Ε, στη χώρα μου τρει φορέ χρειάστηκε να μεταφέρουμε αυτή την οδηγία. Υπάρχουν τρει νόμοι, συνεπώ την εφαρμόζουμε και υπέρ των δέων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μα όπως είπατε κύριε Γιουγκύρος, γιατί ε, είναι πρόβλημα να πληρώσει κανεί περισσότερο. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά η διάταξη όπω έχει συνταχθεί σήμερα δημιουργεί νομικά προβλήματα και πρακτικά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο δεν τη δεχόμαστε. Εάν αποδειχθεί ότι η πρότασή σα είναι κάτι που από νομική άποψη είναι εφαρμόσιμη και από πρακτική άποψη και μπορεί να γίνει δεκτή από τι επιχειρήσει και το καλό των εργαζομένων, τότε τα πράγματα διαφέρουν. Γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω ότι στη μεταλλουργική βιομηχανία αναζητούμε ένα κείμενο το οποίο θα εφαρμόζεται από νομική άποψη και από πρακτική άποψη. Ευχαριστώ. δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα, θα περιοριστώ στα τρία σημεία που έθιξε ο κ. Ουγγέριος και επίσης κατά πόσο είναι ένα πρόβλημα Ανατολής Δύσης. Εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, εάν είναι ένα θέμα Ανατολής Δύσης, εάν δεν απατώμε, το πρόβλημα που αναφέρατε είναι κατά πόσο αυτή η απόσπαση αφορά την έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων. Ναι, γι' αυτό επανήλθα στους ε, ιδρυτικού πατέρε. Αυτό υποτίθεται έπρεπε να κάνει. Και η αγορά θα πρέπει να έχει ισορροπία και όταν υπάρχει έλλειψη εργαζομένων, ορισμένων ειδικοτήτων σε μια χώρα, θα πρέπει να του φέρει από άλλη χώρα. Εάν. Ε, ε, τώρα, περνάμε από τη λειτουργία της οδηγίας από το 1996 μέχρι τώρα, λειτουργεί καλά. Τα προβλήματα προέκυψαν μετά το 2007 και ένα από τα προβλήματα ήταν ότι τα δικαιώματα περιορίζονταν ε, στην εφαρμογή των δικαιωμάτων για τους εργαζομένους, αλλά δημιουργ... επίσης προκαλούσε αθέμητο ανταγωνισμό. Για ορισμένε εταιρείε ε, ήταν... Ε, χρειάζονταν ένα επιχειρησιακό μοντέλο για να στείλουν στη άλλη χώρα εργαζόμενους, επειδή ήταν ευθυνότερη εργασία εκεί. Αυτό όμως δημιούργησε τα προβλήματα. Και γι' αυτό όλη η εσωτερική αγορά αντιμετώπισε ε, πρόβλημα, κυρίως στον οικοδομικό κλάδο. Αντιλαμβάνομαι ότι στον μεταλλουργικό τομέα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το πρόβλημα κατά κλάδων. Στον οικοδομικό τομέα όμω αυτό στρέβλωσε την αγορά. Και όχι μόνο στου εργαζόμενου οι οποίοι είναι αντικείμενο εκμετάλλευση, αλλά και στι εταιρείε. Επειδή το κοινωνικό ντάμπινγκ, αν υπάρχει, σημαίνει εκμετάλλευση των εργαζομένων πρώτον και δεύτερον ανταγωνισμός άνισος κακό για τις εταιρείε, αλλά επίσης σημαίνει φοροδιαφυγή. Όλα αυτά τα στοιχεία σημαίνουν κοινωνικό ντάμπινγκ. Το δεύτερο που αναφέρατε, αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, ναι. Αυτό δεν θα πρέπει να ευθυγραμμίζει όλα τα κοινωνικά μοντέλα στην Ευρώπη. Αυτό είναι εξωρεαλιστικό και αναφερθήκατε στη Δανία, εγώ γνωρίζω την Σουηδία. Αλλά αυτά τα μοντέλα μοιάζουν, νομίζετε. Όχι, δεν μοιάζουν. Δεν μπορεί κανεί να ευθογραμμίσει τα κοινωνικά μοντέλα τη Ευρώπη και δεν θα πρέπει να είναι ο στόχο τη οδηγία. Αλλά υπάρχουν ορισμένε αρχέ που θα πρέπει να θεσπιστούν και αυτέ οι αρχέ είναι να υπάρχει ένα ισότιμο παιχνίδι για τι εταιρείε για του εργαζόμενου. Τώρα, η νομική βάση. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν δεδομένου ότι αυτό δεν αφορά μόνο υπηρεσίες διασυνοριακές, θα πρέπει να υπάρχει διεύρυνση τη νομική βάσης, επειδή η συνθήκη μα έχει αλλάξει σε σχέση με το 96. Τέλος, κατά πόσο είναι πρόβλημα ανατολή Δύση. Δεν το νομίζω. Δεν θα έπρεπε, διότι θα ήταν πρόβλημα ανατολή Δύση, εάν θεωρούσαμε την απόσπαση μόνον ένα μέσο για να έχουμε χαμηλότερο εργατικό κόστος ενώ όπως αναφέρθηκε <clears throat> σχετικά με την έλλειψη ε, ειδικοτήκων σε μια χώρα και το θέμα της ισότητας, της, ε, ε, της δικαιοσύνης και η αποτελεσματική χρήση της αγοράς δεν είναι πρόβλημα το Ορισμένες χώρες ε, πάντοτε είχαν το πρόβλημα κατά πόσον πρέπει να δίνουν ίση αμοιβή για ίση εργασία. Αυτό ήταν πρόβλημα στη Σουηδία, στη Γερμανία και το ζητούμενο είναι ότι ε, κατά πόσο το κράτος μέλος που το κάνει αυτό ε, έχει και μια πιο αποτελεσματική οικονομία, μια μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη ανάπτυξη και οι χώρες που στηρίχτηκαν σε στρατηγικές χαμηλότερου κόστους αυτό ακολούθησαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Πάτρικ Κλέμπους έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Μιλήσαμε για μία μελέτη. Ο κύριος Μπανιό είπε ότι 16 επιχειρήσεις <coughs> συμμετείχαν. είναι δυνατόν να αναφερθούμε μόνο σε 16 επιχειρήσεις. Στη Γαλλία υπάρχει μια δίκη αυτή την εποχή για μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία. Ξεκίνησε χτες και συνεχίζεται σήμερα. 3.000 άτομα εργαζόταν σε ένα εργοτάξιο και 460 επιτόπου, εκ των οποίων οι 295 ήταν με παράνομες συμβάσεις στη Γαλλία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε για ασφάλεια. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες είναι θύματα εκμετάλλευσης και εκμεταλλεύονται κάποιους άλλους με τη σειρά τους. Και βεβαίως ξέρουμε ότι οι συμβάσεις αυτές βασίζονται σε κανόνες οι οποίοι είναι καθαρά καταναγκαστικοί. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να διακόψει, να διακοπεί μάλλον η σχέση εργασίας τους και να ξανασταλεί στη χώρα του από τη μία μέρα στην άλλη. Πρόκειται για την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Μυθιστορήματα έχουν γραφτεί γι' αυτό το φαινόμενο και είναι σκανδαλώδες το ότι σήμερα αυτή η απάνθρωπη μεταχείριση συνεχίζεται. Και αυτό ισχύει και για τις συνθήκε εργασίας και για τις συνθήκε διαβίωσης και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που τουλάχιστον ξεκινάει αυτή η συζήτηση, γιατί κάποια πράγματα θα ακουστούν, θα γραφτούν και ενδεχομένως μπορεί να βρούμε και κάποιες λύσεις. Για να υπάρχει εδώ ασφάλεια στις επιχειρήσεις και εδώ εκπροσωπώ μεσές και μικρομεσές επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκοβών. Σήμερα είμαι βιοτέχνης. Προηγουμένως όμως ήμουν εργαζόμενος, υπάλληλο σε ένα μεγάλο όμιλο. Γνωρίζω λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει. Η κυρία Μογά Σαχτιέ αναφέρθηκε και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, στην μαθητεία και στην συνεχή και διαβίου κατάρτιση. Εάν υπήρχαν τέτοιου είδους προβλέψεις, θα είχαμε αποφύγει πολλά από αυτά τα φαινόμενα. Στη Γαλλία υπήρχαν πάνω από 26.000 αποσπασμένοι εργαζόμενοι το 2004 και συνεχίζουμε να έχουμε περίπου τον ίδιο αριθμό αποσπασμένων και 6 εκατομμύρια άνεργους. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε αυτούς τις 6 εκατομμύρια άνεργους να μην βρίσκουμε εργαζόμενους για να μπορούν να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Θα πρέπει ίσως να δούμε τα πραγματικά αίτια αυτών των αποσπάσεων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Επαναλαμβάνω το αίτημά μου. Αν μπορείτε να στείλετε τις παρουσιάσεις σας καθώς και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις στις οποίες δεν προλάβατε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ <coughs> όλους σας και η γραμματεία θα έρθει σε επαφή μαζί σας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε με την εισηγήτρια, με τις δύο εισηγήτριες, την κυρία Μογάν Σαντιέ και την κυρία Αγκάριος. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των εμπειρογνωμόνων μας που μας έδωσαν τις θέσεις και τις αναλύσεις τους και τις διάφορες απόψεις τους. Να απαντήσω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, μιας και μιλήσαμε για την εκτελεστική πράξη της οδηγίας και τι γίνεται με αυτήν. Να επενθυμίσω ότι οι δύο συνηγήτριες, οι συγήτριες, οι Αγνές και εγώ, θα γράψουμε μια κοινή επιστολή στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, Σλοβακία δηλαδή, στον Σλοβάκο Πρωθυπουργό, για να ζητήσουμε ακριβώς την εφαρμογή της οδηγίας που η κυρία Ζογιέσκα προετοίμασε τον Απρίλιο του 2014. Εμείς λοιπόν ήδη έχουμε κινητοποιηθεί για αυτό το θέμα. Αλλά πέραν τούτου θέλουμε να δείξουμε στο Συμβούλιο ότι εμείς χρειαζόμαστε αυτή την εκκλαστική οδηγία. Όμως δεν είναι αυτό το αντικείμενο της αναθεώρησης της οδηγίας για τους ε, αποσπασμένους ένα κείμενο δεν αντικαθιστά το άλλο. Θα πρέπει και τα δύο να εκτελεστούν. Και πάνω στα δύο θα πρέπει να δουλέψουμε. Ιδιαίτερα για τα θέματα των αμοιβών, των ορισμών των αμοιβών. Τι εννοούμε με τον όρο αμοιβή και ποια είναι η διάρκεια της απόσπασης. Πώς θα πρέπει αυτά τα γραφεία νοικίασης εργαζομένων να εργαστούν ώστε να μην εκμεταλλεύονται τα ίδια αυτά τα γραφεία τους αποσπασμένους εργαζόμενους, υπεργολαβία και συλλογικέ συμβάσεις. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα για τα οποία ήδη έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι αποσπασμένοι να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης πανευρωπαϊκά με ένα σαφές και εφαρμόσιμο και εποπτεύσιμο κείμενο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ελιζαμπέτ. Τώρα, Αγνές, η σειρά σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ και που μοιράζομαι τις σκέψεις μου μαζί σας. και πέρα από τόσο είπε η συνεισηγήτριά μου, θα ήθελα να κάνω και εγώ έκκληση σε εσά. Επειδή αυτή η ακρόαση έγινε στη σωστή στιγμή, επειδή τώρα ετοιμάζομαι την απάντησή μας στην πρόταση της Επιτροπής. Και νομίζω ότι το είπα πρωτήτερα, κατηδίαν σε ορισμένα άτομα και έχω γράψει και μια επιστολή από αυτού σε ορισμένα άτομα μεταξύ των εμπειρογνωμόνων μας. Θα ήθελα να σας πω το εξή. Εάν θέλετε τελικά να έχετε μία εφαρμόσιμη πρόταση, να μας βοηθήσετε χρησιμοποιώντας την εμπειρία σας ώστε να μας κάνετε και εσείς συγκεκριμένες προτάσεις. Διότι νομίζω ότι είναι σημαντικό η τελική διατύπωση να αντικατοπτρίζει αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της παροχής υπηρεσιών, αλλά το επαναλαμβάνω και την ελευθερία να μην είναι κανείς αντικείμενο εκμετάλλευσης στην διαδικασία αυτή. Και επίσης είναι σημαντικό να μην υπάρχει εκμετάλλευση των ατόμων και τα άτομα στην αγορά εργασίας να καλωσορίζουν και τους νέους μετανάστες που έρχονται σε αυτή την αγορά, αλλά να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση των ατόμων. Και χαιρετίζω το γεγονός ότι μετά από αυτή την ακρόαση, όχι μόνον είδαμε ποια είναι τα προβλήματα που επισημάνθηκαν, αλλά Ορισμένοι μας είπαν ότι θέλουν να βοηθήσουν για να επιληθούν σωστά αυτά τα προβλήματα. Επειδή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι σημαντικό το project αυτό να είναι ισορροπημένο ανάμεσα δηλαδή την ελευθερία της παροχής υπηρεσιών και την προστασία των εργαζομένων. Όχι μόνο οι εργαζόμενοι που στέλνονται στο εξωτερικό σε απόσπαση, αλλά και εκείνοι που υποδέχονται τους νέους συναδέλφους. Αυτή λοιπόν η εξισορρόπηση γίνεται πρώτα από εμά. Αλλά χρειαζόμαστε και τη δική σας τη βοήθεια, την οποία εκτιμούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή είναι παρούσα εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον η Επιτροπή επιθυμεί να αντιδράσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, στη συντομία θα ήθελα να σας πω ότι παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις. Θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω ότι η οδηγία 96-71 δεν είναι η οδηγία που θεσπίζει την ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών που προβλέπεται από τη συνθήκη, αλλά οδηγία η οποία προβλέπει προστασία των αποσπασμένων. Γι' αυτό πρέπει να έχετε υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας πρέπει να παραμείνει για να προστατευθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε από πολλούς εδώ. Και θα ήθελα απλώς να το υπογραμμίσω. Εξάλλου, το κεντρικό θέμα το οποίο προέκυψε είναι κατά πόσον αυτή η οδηγία προστατεύει πάντοτε επαρκώς ε, τους εργαζόμενους αυτούς. Δύο θέματα αναφέρθηκαν. Η υλοποίηση και η καταπολέμηση κατά των καταχρήσεων και ήθελα να το επιβεβαιώσω. Η Επιτροπή αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην υλοποίηση της οδηγίας 2014-67 η διαδικασία παρεμβάσεων έχει ξεκινήσει κατά των χωρών που δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία και ε, εξετάζουμε αυτά τα μέτρα μεταφοράς ε, με αυστηρό τρόπο. Το δεύτερο το οποίο συζητήθηκε εδώ είναι η εφαρμογή των βασικών κανόνων της οδηγίας και κατά πόσον ε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αναβάθμιση της οδηγίας μετά από 20 χρόνια σε σχέση με πιο πρόσφατα έγγραφα, κυρίως την προσωρινή εργασία ή για τη μακροχρόνια απόσπαση που μπορεί να ενσωματωθεί στην κοινωνική ασφάλιση και αφετέρου υπάρχουν κανόνες οι οποίοι πρέπει να είναι δίκαιοι. Δηλαδή ότι υπάρχουν ήδη κανόνες που θα εφαρμόζονται στις τοπικές επιχειρήσεις και στις αποσπασμένες επιχειρήσεις όταν παρέχουν υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you all of you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και τις εισηγήτριες και τους σκιώδεις. Δεν είναι εύκολο θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα βρεθούν λύσεις ικανοποιητικές για όλους μας. Ευχαριστώ και τους Γερμηνείς. Meeting. Επόμενη συνεδρίαση. Συγγνώμη, ξέχασα. Όχι, το επόμενο θέμα. είναι τα διάφορα. Δεν υπάρχουν όμως διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 29 Νοεμβρίου από τις 9 ως τις 6.30. Εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ.